Έχουμε. Ε, το ψήσμα για την Γουνέα Συμφωνία Μερμεσία Διάταξη. Ο κ. Ματσάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ιουνέα έχει γνωρίσει μια πολύ τάραχη ιστορία, διότι έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συνεχώς εμπλέκονται στην ιστορία της κατά το παρελθόν. Το 15ο ανακατακτήθηκε από την Πορτογαλία και ε, χρεώθησαν να γίνουν σκλάβοι με το ευρωπαϊκό δουλεμπόριο. Το 1880 επικίστηκε από τη Γαλλία το 1958 επέκταση ανεξαρτησία συνδέθηκε με τη Σοβιετική Ένωση και η μεταπιοκρατική ιστορία τη χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτισμό. Η δε αρχηγοί αυτή τη χώρα ε, κυβερνούν βασιζόμενοι στον πρωτόγνωρο στρατό. Έχει αλουμίνιο, ε, διαμάντια, χρυσό και ουράνιο. Είναι μία από τι πιο φτωχέ χώρε του κόσμου. Αυτό ο πλούτο τη χώρα γίνεται αντικείμενο από Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά. Ε, Επίση υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στα πλαίσια της ε, διακυβέρνησης της χώρας και οι εταιρείε φυσικά δεν ενδιαφέρονται για την ευημερία των ε, πολιτών και οι διαμαρτυρίες των ανθρώπινων δικαιώματα ξεκίνησαν μόνο όταν κινδυνεύουν τα οικονομικά δικαιώματα της αργούσας τάξης. Έχει τώρα λοιπόν κάποιον δικτάτορα ε, και είναι ένας, λέγεται Καμάρα, είναι ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος ε, είναι επικεφαλής αυτής της διαφθοράς ε, και έτσι τα 10 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας δεν μπορούν να φτάσουν μια κατάσταση ευημερίας. Δεν έχω ιδέα κατά πόσον πραγματικά αυτά τα οποία εξαγγείλει για βελτίωση κατάσταση του λογαγός Καμάρα θα τα κάνει και αν τα θέλει πραγματικά. Πάντως, τι ε, τελευταίε δεκαετίε το να τόσο άσχημο που δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Η δε Ευρώπη αλλά και ο υπόλοιπο κόσμο, με σταυρωμένα τα χέρια παρακολουθεί το πώ ο ορυκτό πλούτο τη χώρα γίνεται κειμένο Ε, βλέπουμε επομένω ότι πρόκειται και εδώ για μια στρατική δικτατορία και έτσι καλώ είναι κάτι κακό και ελπίζουμε να γίνει μετασχηματισμό δημοκρατικό κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ματσάκη. Ο Ντίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σοντή, αγαπητέ Επίτροπε, κύριε Σπίτλ, αγαπητοί συνάδελφοι. Στι 22 Δεκάτου του 2008 ο Πρόεδρο εξαφανίστηκε ε, το 1974 μέσα σε μια νύχτα 22 Δεκεμβρίου. Ε, έγινε τότε η αλλαγή στην ε, εξουσία με ένα πραξικόπημα. Αυτοί οι επόμενε τώρα που ηγούνται της χώρας χαρακτηρίζονται από του πιο διεφθαρμένου από το Transparency International. Σε αυτή τη πάντως ποτέ δεν υπήρξε κράτος δικαίου και δημοκρατία. 24 ετών είναι ε, ο σημερινός ηγέτης. Ε, το 1958 ήταν ο Σέκο Τουρέ, το, το κατόπιν μαρξιστής και τώρα έχουμε έναν ε, απλό αξιωματικό που ανέλαβε τα ενία της χώρας, ασχολούνταν πριν με, τα, με τις προμήθειες του στρατού, και τώρα έχει εξαγγείλει ότι θα πάει προς δημοκρατία και κράτος δικαίου. Και επίσης, όπως για το Σύνταγμα, θα πάει για εκλογές. Στις 24 Δεκεμβρίου αυτός ο άγνωστος ε, λοχαγός, αυτόν εγκαιρίχθηκε πρόεδρος, ε, χιλιάδες κόσμου τον ε, χειροκρότησαν και ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας έτσι με τρόπο τελεσυγραφικό αποφάσισε να γίνουν εκλογέ το 2010, να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ε, έχει επίσης πρωθυπουργό κάποιον ε, διπλωμάτη και τώρα προσπαθεί να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και με την αντιπολίτευση. Βεβαίως και θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτό το πραξικόπημα και αυτό κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα. Βεβαίω και χρειάζονται πολιτικέ λύσει για να βγει καμία σε μια διατορία. Τα πράγματα δεν είναι ε, απλά. Επομένω, εμεί προτείνουμε να εγκριθεί αυτό το ψήφισμα. Σα ευχαριστώ και τώρα για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριο Μάιερ. Το 2007, το Φεβρουάριο, συζητήθηκε εδώ ένα κατεπήγον ψήφισμα το οποίο αφορούσε την δικτατορία του κυρίου Λασανά, ο οποίος από το 1994 ήταν στο πηδάλιο της χώρας και συνεπεριφέρεται ε, σαν ήταν ιδιοκτησία του η χώρα όλα τα πολιτικά κόμματα ήταν κατά αυτών εκλογών που αυτός εξήγηλε και δεν επίσημη θέση ε, των κομμάτων ήταν να εγκαταλείψουν το κοινοβούλιο καταστολή ακολούθησε. Το 2007 είχαμε 59 νεκρούς σε κάποιο ε, σελτήριο το οποίο έγινε και ε, το Δεκέμβριο του 2008 είχαμε αυτό το πραξικόπημα το απροσδόκητο οπότε άλλος πήγε στην εξουσία και δεν ξέρουμε τώρα αν θα υπάρξει δημοκρατική αλλαγή. Δεν ξέρουμε εάν τώρα θα έχουμε αλλαγή ή εάν θα έχουμε έναν νέο δικτάτορα ο οποίος ε, θα ενδιαφέρεται για πλουτίσια από τους πόρους της χώρας και Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί αφρικανικοί φορείς έχουν καταδικάσει αυτό το πραξικόπημα. Γαλλία, Σενεγάλη ζητούν την προκήρυξη εκλογών μέσα στο διάστημα του ενός έτους. Άρα θα πρέπει να ακούσουμε την αντιπολίτευση που είπαμε ότι έχει αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο και στο περιθώριο θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί ο λαός της χώρας και θα πρέπει η χώρα να διηγηθεί σύντομα σε εκλογές. Δεν χρειάζεται καινούργιο δικτάτορα η χώρα. Χρειάζεται με μια δημοκρατική αλλαγή ταχαίως. Κούσμακα. Κάσμαρ, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Στη Δυτική Αφρική φαίνεται ότι τα πραξικοπήματα ήταν ο μόνος τρόπος να διεκδικήσουν την εξουσία και στη Σιέρα Λεόνε, στην ακτή του Ελεφαντοστού, στη Σιέρα Λεόνε και στη Λιβερία επήλθαν πολιτικές αλλαγές, ε, γεννήθηκαν νέες δημοκρατίες, ενώ η Γουινέα έχει μείνει σε αυτό το παρελθόν. Ο πρώην πρόεδρος κ. Κοντέ, που έγινε και αυτός πρόεδρος ε, μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος, ε, ήταν μόλις ο δεύτερος πρόεδρος ε, της Γουινέας θα πρέπει η περαιτέρω βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Γουινέα να εξαρτηθεί από την αποκατάσταση τη ε, ειρήνη και τη Δημοκρατία και από τη διεξαγωγή εκλογών. Και η σωστή διεξαγωγή των εκλογών θα πρέπει να επιτηρείται από διεθνεί ε, οργανισμού. Εάν ο κύριος ε, να θέλει να γίνει ο Ομπάμα τη Δυτική Αφρική, θα πρέπει να αλλάξει η διαφθορά και η φτώχεια. Ευχαριστώ κυρία Τομασέφσκα. Δύο λεπτά για την Ευρώπη των Εθνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Μία μέρα μετά το θάνατο του Προέδρου Λενθάνα Κοντές στις 23 Δεκεμβρίου 2008 η στρατιωτική Χούντα ανέλαβε το καθεστώς ε, και διέλυσε την ε, κυβέρνηση της χώρας. Οι εκλογές πρόκειται να γίνουν το 2010, ενώ θα έπρεπε να οργανωθεί κάτι μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Η Αφρικανική Ένωση διέκοψε, ανέστηλε ε, την ιδιότητα μέλους της Γουινέας και νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να ζητήσει να γίνουν δημοκρατικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε ότι θα δώσει ανθρωπιστική βοήθεια και για να υποστηρίξει τους πολίτες και να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο με τις αρχές. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω τέσσερις εγγεγραμμένους. Σε δύο μπορώ να δώσω το λόγο, αλλά αν τηρήσετε το χρόνο σας, μπορεί να μιλήσετε και όλοι. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος Λανσάνα Κοντέ ήταν το αρχέτυπο ενό του ισχυρού αφρικανικού άνδρα διεφθαρμένος που κυβερνούσε τη χώρα με σιδερένια γροθιά. Ο θάνατος του Κοντέ προσέφερε μια ευκαιρία στην, ε, στην Γουινέα να γυρίσει σελίδα στην ιστορία της. Ε, βέβαια, οι, οι, οι ελπίδες αυτές για πραγματική δημοκρατία διαψεύστηκαν από το ε, πραξικόπημα. Δεν, βέβαια, η χούντα αυτή προφανώς δεν μπορεί να ληφθεί ε, σοβαρά υπόψη από την ε, διεθνή κοινή γνώμη και την ε, διεθνή κοινότητα εν γέννη, εάν, δεν, αν καθυστερούν και δεν κάνουν κάτι σημαντικό. νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να περάσουμε στην διαδικασία των ακυρώσεων. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε, θα πρέπει μάλλον να, να, απαιτήσουμε μέσα στα πλαίσια των, συμφωνιών μας ε, να διασφαλιστούν κάποια δημοκρατικά, βασικά δημοκρατικά δικαιώματα σε αντάλλαγμα με τις εμπορικές ε, σχέσεις. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. mamy kolejny przypadek gdzie ναι. Πρόεδρε, αυτή η δικτατορία ακολουθεί με προβλέψιμο τρόπο. Πρώτα πρώτα να στέλνουν το Σύνταγμα και κατόπιν υπόσχονται δημοκρατικές εκλογές. Λένε για μια περίοδο διετίας αλλά σύντομα αυτό που γίνεται, αυτοί όλοι οι αξιωματικοί βρίσκουν θέση στην κυβέρνηση και πάμε προ παραβιάσει ε, δημοκρατικών αρχών, καταστολή, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι ελπίζουμε ότι ίσω, ίσω ανακύψει κάποια λύση, ίσω έχουμε διαφορετικό σενάριο από τα πάγια. Πάντω δυστυχώ ε, το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να ασκήσουμε κάποια πίεση είναι εάν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε η Ένωση Δυτικής Αφρικής που αποφάσισε να αναστείλει τη σχέση με τη χώρα να τις διακόψει. Ξέρουμε ότι συνέχεια μειώνει το κατεφαλήν εισόδημα. Άρα θα πρέπει να δείξει ποινή η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσει ότι θα επανέλθει στους μαλλούς ρυθμούς η δημόσια ζωή της χώρας για το καλό του λαού της. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μιλούμε για την Γουινέα, μια χώρα που σήμερα με το Transparency International είναι από τις πιο διεφθαρμένες στην Αφρική. Τα στοιχειώδη, τα χρειώδη δεν έχει και ο κόσμος ζει σε τραγικές συνθήκες. Ε, πρόκειται για κάποιο πλήρως παράνομο πραξικόπημα και βλέπουμε ότι έχει ολόκληρη παράδοση σε τέτοια ε, πραξικοπήματα η χώρα. Δεν έγιναν τελικά εκλογές όπως θα όφελαν να γίνουν πρώτα μια διορία. Άρα χτυπάει το καμπάνι του συναγερμού για τη διεθνή κοινότητα. Για όποια χώρα και αν επρόκειτο θα είχαμε αστάθεια, θα είχαμε αιματοχυσία. Επομένως, να περάσει το ψήφισμά μας και να ζητήσουμε έτσι εκλογές σύμφωνα με τα αποδεκτά διεθνώς πρότυπα, σύμφωνα με τους διεθνείς φορείς της, της Δυτικής Αφρικής. Και να υπάρξει και παρατήρηση των εκλογών, για αλλιώς θα πρόκειται για μια φάρσα. Ο επόμενος, κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτό το πραξικόπημα στη Δυτική Γουινέα. Και εδώ το σενάριο ήταν προβλέψιμο όπως έχει γίνει και αλλού στην Αφρική ή και σε άλλες επίρους. Και πριν από 24 χρόνια με παρόμοιες πρωταγωνιστές είχαν γίνει τα ίδια αν λήφθη μόνο στρατιωτική δράση ε, και οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την, ε, τις κυβερνητικές θέσεις. Η ΔΕ Αφρικανική Ένωση ανέστηλε διπλωματικές χώρες με την χώρα εκείνη. Συμφωνώ δε ότι πίεση από έξω μπορεί να αποδώσει κάποια αποτελέσματα και ίσως πρόξει χώρα προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουν δημοσιευτεί κάποιες κάποιε προτάσει από τι ευρωπαϊκέ χώρε, σύμφωνα με τι οποίε ίσω ε, μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οπότε και εμεί προτείνουμε να επιψηφιστεί το κείμενο. Κύριε Σπίτλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Οι ειδήσει ε, σχετικά με το θάνατο του Προέδρου της Γουινέας Λανσάνα Κοντές στις 22 Δεκεμβρίου του 2008 ακολουθήθηκαν στη συνέχεια από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα και διάλυση των δημοκρατικών των θεσμών του κράτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη δήλωση του Συμβουλίου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγγέλει αυτό το πραξικόπημα και ζητούμε από τη χώρα να επανέλθει στην ε, μη στρατιωτική διακυβέρνηση. Είναι σαφές ότι οι συνθήκες διαβίωσης ε, για τους πολίτες της Γουινέας είναι τόσο κακές που ακόμη και ένα στρατιωτικό πραξικόπημα μπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη, κάτι το οποίο μπορεί να φέρει την υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλος, μέλλον. Επίσης, αυτό δείχνει ότι το προηγούμενο καθεστώς στη χώρα είχε χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη του σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που οι πολίτες προτίμησαν το στρατό που ανέλαβε την εξουσία ε, έναντι των ε, συνταγματικά υποτίθεται εκλεγμένων εκπροσώπων. Χρειάζονται αποτελεσματικές ε, και γρήγορες κινήσεις από τη διεθνή κοινότητα. Ο κύριος Τσάμπας, πρόεδρος της ΕΚΟΒΑΣ, της Οικονομικής Ένωσης Χωρών της Δυτικής Αφρικής, και η Ένωση Χωρών της Δυτικής Αφρικής ανέστηλαν την ιδιότητα μέλους της Γουινέας και κατήγγυλαν το πραξικόπημα. Η Επιτροπή προτίθεται να ακολουθεί τις προσπάθειες που καταβάλει η ΕΚΟΒΑΣ ούτως ώστε να επιταχύνουμε την επάνωδο της Γουινέας σε ένα καθεστώς όπου θα ε, διοργανωθούν δημοκρατικές εκλογές και η πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα είναι το πώς θα μπορέσει να υποστηρίξει τη Γουινέα στη μετάβασή της στη δημοκρατία και στην οργάνωση ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών για, το νομοθετικό τους, ε, για την νομοθετική του συνέλευση και για τον πρόεδρό του. Το Μάρτιο του 2004, μετά από εκλογές οι οποίες δεν σέβονταν τις αρχές της δημοκρατίας και παραβίαζαν σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού, αποφασίσαμε να αρχίσουμε διαβουλεύσεις μεταξύ Γουινέα ε, και Ευρωπαϊκής ένωση σύμφωνα με το άρθρο 96 τη Συμφωνία Κοτονού επιτύχαμε πρόοδο στου εξή τομείς. Δημοτικές εκλογές το 2006, απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης, αναθεώρηση του εκλογικού πλαισίου από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και βελτίωση του μακροοικονομικού πλαισίου. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαδικασία των εκλογών που άρχισε ε, πέρυσι τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί και την ε, Τετάρτη μια κοινή αποστολή Προεδρίας και Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεταβεί στη Γουινέα. Υποστηρίζουμε πολλές από τις κινήσεις της ΕΚΟΒΑΣ και της ε, Ένωσης των χωρών της Δυτικής Αφρικής και θέλουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση στη χώρα και να προτείνουμε μέτρα τα οποία θα υποστηρίξουν τη Γουινέα στη μετάβασή της στη δημοκρατία. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Σε 20 λεπτά περίπου, στο τέλος των απογευματινών μας συζητήσεων, θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα. Τώρα έχουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος ε, για την ελευθερία του τύπου στην Κένια. Τον λόγο τον έχει ο κύριος Ματσάκης, σαν συντάκτης της, ε, του ψηφίσματος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ελευθερία του τύπου ε, είναι ταυτόσιμη με την ελευθερία έκφρασης. Αυτό βέβαια δεν εφαρμόζεται στην ιδανική, ιδανικά σε, στην δική μας